Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε την κοινή συνεδρία των τριών επιτροπών μας. Της Επιτροπής Εξωτερικών Ανάπτυξης και Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους σας. Ας ξεκινήσουμε παρακαλώ αυτή την κοινή μας συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Νιώθω μεγάλη τιμή που συμπροεδρεύω μαζί με τις συναδέλφους ε, Λίντα Μακάβαν, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης και την κυρία Ελένα Βαλενσιάνο, που είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμπροεδρεύουμε αυτή την ε, συνεδρίαση που, που ε, διοργανώνουμε ε, μία φορά το έτος με τους βραβευθέντες με το ζαβείο, βραβείο Ζαχάροφ. Και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα σήμερα την κυρία Νάντια Μουράντ, και την κυρία Λάμια Χάτζι Μπασάρ, που είναι οι δύο βραβευτήσεις με το βραβείο Ζαχάροφ του 2016. Θα ήθελα επίσης ε, να καλωσορίσω και δύο άλλους υποψηφίους που ήταν και οι φιναλίστ, τον κύριο Μουσταφά Τζεμίλεφ και τον Τζαν Ντιντάρ που έπρεπε κανονικά να έρθει, αλλά δυστυχώς κάποια προβλήματα οργανωτικά και ευελπιστούμε ότι θα καταθάσει αργότερα. Ο κύριο Τζεμίλευ, έχετε και μετάφραση διερμηνή από τα ρωσικά, μπορείτε αν θέλετε να μιλήσετε. Ε, και θα έχετε την ευκαιρία προς το τέλος συνεδρίασης να κάνετε και εσείς μια σύντομη παρέμβαση. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον συνάδελφο David Campbell Bannerman, που είναι πρόεδρος αντιπροσωπείας μας για τις σχέσεις με το Ιράκ, ε, τη χώρα από την οποία ε, κατάγονται οι δύο ευρωπευθύσεις μας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει το βραβείο Ζαχάροφ για την ε, ελευθερία σκέψης από το 1988 σε άτομα ή οργανώσεις που με τις δράσεις, σκέψεις και μαρτυρίες τους μας υπενθυμίζουν πόσο απαραίτητο είναι για το δημοκρατικό βίο μιας χώρας να σέβεται και να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και στα χρόνια αυτά το βραβείο Ζαχάροφ έχει γίνει από τις πιο απτές εκφάνσεις της συλλογικής διακομματικής δέσμευσής μας υπέρ της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της στήριξής μας και της συμπαράστασής μας με εκείνους που δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους υπέρ της ελευθερίας και της δικαιοσύνης στον κόσμο. Σε πολλά μέρη του κόσμου ακόμη Άτομα και ομάδε εξακολουθούν να δίνουν καθημερινά τη μάχη του για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δυνατότητά του να λαμβάνουν τι αποφάσει του και να καθορίζουν τη ζωή και το μέλλον του. Αυτό ο συνεχή αγώνα σε πολλά μέρη του κόσμου μα δείχνει πόσο ανεκτήμητο και σπουδαίο είναι αυτό το πλαίσιο και πόσο εύκολα μπορεί να συντριβεί. Στου χαλεπού καιρού που βιώνουμε και ενώ περνούμε από τη μια κρίση στην άλλη, με μαζικέ ισορές προσφύγων και με την πρόκληση τη τρομοκρατία, δεν θα πρέπει να δώσουμε στο πειρασμό να διακυβεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα που πασχίσαμε να υλοποιήσουμε ε, και να μην τα θυσιάσουμε στο βωμό τη περισσότερη απλώς ασφάλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα τιμούμε του βραβευθήσεις με το βραβείο Ζαχάροφ, την δεσπινίδα Νάντια Μουράντ και τη δεσπινίδα Λάμια Χατζή Μπασάρ, και μαζί τους θυμούμε και όλους εκείνους τους ανθρώπους που παλεύουν και αγωνίζονται καθημερινά στις τοπικές κοινότητες ή ε, διεθνώς για να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, χωρώντας τους έτσι την οικουμενική τους αξία. Θα ήθελα επίσης να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφό μου, την κυρία Ελένα Βαλενσιάνο, που είναι πρόεδρος Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρακαλώ, Ελένα, έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους και όλες που ήρθατε απόψε για να μπορέσουμε να είμαστε με δύο ξεχωριστές γυναίκες που το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι είναι οι νικήτριες του διαγωνισμού για το Ραδιοζάχος 2016. Εκεί που μία μικρή ε, κοινότητα δίνει τη μάχη της στα βουνά της Τουρκίας. Πάνω από 4.000 χρόνια ιστορία έχει αυτός ο λαός και πάντοτε υφίστανται διώξεις και άλλη μια φορά έχουμε μια μαύρη ιστορίας βάρος αυτών είναι οι πρώτοι που υπέστησαν τον 21ο αιώνα γενοκτονία και το Ισλαμικό κράτος εγκατέστησε με κάποια πρόφαση θρησκευτική αυτό το κράτος τρόμου στην περιοχή. Κάρλα. Οπότε βλέπουμε τώρα το πώς υποφέρουν οι Γεζιντοί και αυτό γίνεται από κάποιες φωνές όπως της ε, Λαμία και όπως της Νάντια. Και αυτές τις ε, πήραν από την ε, ελληνική ζωή τους, τους ξερίζωσαν και αυτές από τότε αυτό το οποίο πέρασαν είναι κάτι το απερίγραπτο και είναι σαν να μην υπάρχουν πια αυτές και οικογένειά τους γιατί υπέστησαν βασανιστήρια, βασανιστήρια σωματικά και ψυχολογικά ε, τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν το ότι πέρασαν εδώ είναι όμως και κατάφεραν να ξεφύγουν κατάφεραν να φτάσουν μέχρι την Ευρώπη και κατάφεραν να σηκώσουν κεφάλι Οπότε το βραβείο δεν είναι για τα όσα περάσαν, είναι για το θάρρος τους. Ούτε επίσης για το ότι πέρασαν ε, σεξουαλική δολία από πλευράς των τζιχαντιστών, αλλά και κατάφεραν να το ξεπεράσουν. Και αναγνωρίζουμε το θάρρος αυτών των ε, δύο γυναικών. Αυτό το κάνουμε και στο όνομα όλων των χιλιάδων άλλων γυναικών που συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τον ζυγό του Ισλαμικού κράτους στη Βόρεια Συρία και να υποφέρουν ε, αφάνταστη βία. Οπότε το να βοηθήσουμε αυτές τις πιο ευάλωτες, αυτές που έχουν διωχθεί περισσότερο, τις πιο ξεχασμένες. Αυτός είναι ο στόχος του βραβείου Ζαχάροφ φέτος. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό το οποίο ε, αισθάνεται τιμή του να μπορεί να δώσει αυτό το βραβείο Ζαχάροφ στην ε, Λάμια και στην Άντια, γιατί βρήκαν τη δύναμη να δώσουν αυτόν τον αγώνα για την οικογένειά τους, για το λαό τους, για τις ε, συντροφισές τους και για όλες τις άλλες για όλους που είμαστε εδώ. Αυτό είναι ένα μάθημα αξιοπρέπειας και θάρρος. Οπότε όλοι και όλες θα πρέπει αυτό το μήνυμα, αυτή η φωνή αυτών των γυναικών που μπόρεσαν να ξεπεράσουν τραύματα και φόβους να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. Ούτω ώστε ποτέ καμία άλλη γυναίκα να μην περάσει αυτά τα οποία περάσανε εκείνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας θυμήσατε τι έγινε και γιατί ε, βραβεύσαμε τις δύο κυρίες. Θέλω να πω και στις δύο ότι απονέμετε το βραβείο από το Κοινοβούλιο σε εσά γιατί ο αγώνας σας ήταν σκληρός και είμαστε στο πλευρό σας στον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, χωρίς άλλη καθυστέρηση έχω την τιμή να σας δώσω το λόγο για να, απευθύνετε, να απευθυνθείτε στις επιτροπές μας. Ποιος, ποια κυρία θα μιλήσει ε, πρώτη, κυρία Μουράκη ή η κυρία Μπασάρ. κυρια Μπασάρα, Λαμία Χατζή Μπασάρ. Uh, I thank you very much uh, that you... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το βραβείο με το οποίο μας τιμήσατε. Uh, this shows that... Το βραβείο αυτό δείχνει ότι μας συμπαρίσταστε, μας, μας στηρίζετε, στέκεστε στο πλευρό μας και προσπαθείτε να μας βοηθήσετε και ελπίζω να ενισχύσετε την υποστήριξή σας προς την κοινότητά μας, γιατί έχουμε ακόμη 3.500 γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται εχμάλωτες ακόμη στα χέρια του Νταέσ. Η κοινότητά μας χρειάζεται την θέσπιση μιας διεθνούς ε, ζώνης προστασίας. Και εμείς, η χριστιανική κοινότητα στο Ιράκ, αλλά και άλλες μειονότητες χρειάζονται ε, ασφαλείς ζώνες και χωρίς τη δημιουργία τέτοιων ασφαλών ζωνών και χωρίς ειδική υποστήριξη δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στα εδάφη και στις αιστείες μας. Uh, uh, δεν θα μπορέσουμε να γυρίσουμε στην πατρίδα μας χωρίς αυτή τη βοήθεια γιατί ε, η κοινότητά μας πρόκειται να έχει σφαγή, πρόκειται να έχουν γίνει σκλάβες, να έχουν βιαστεί οι γυναίκες και τα παιδιά α, Αυτά χωρίς τη βοήθεια για την κοινότητα. بهزارە کەچێ دووەکەم هەینە نەبەس ئەزم و هەکە نادیار تنێ بهزارە دووەکەمە هەینە εγώ είμαι μία από αυτές τις ε, Yazidi που έπεσαν θύματα του Ισλαμικού κράτους. Υπάρχουν όμως χιλιάδες από κορίτσια σαν την Αγία, σαν και εμένα, που έπεσαν θύματα ε, αυτών των ε, τρομοκρατών. Υπάρχουν The Zakharov uh, Prize is a... Το βραβείο Ζαχάροφ μας δίνει δύναμη και στις δύο. Αλλά δεν πρέπει να πληθύνεται μόνο σε εμάς τις δύο. Θα πρέπει να πάει σε όλες τις γυναίκες που έπεσαν θύματα του Ισλαμικού κράτους. Ε, uh, another point I want to mention that... Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Μετά την απελευθέρωση του Σιγκάλ κανείς δεν νοιάστηκε για τη σφαγή όλων αυτών. I thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βραβείο αλλά ελπίζουμε ότι θα βοηθήσετε και την κοινότητά μα. Ε, Οι γυναίκε και τα παιδιά που επέζησαν από το Ισλαμικό κράτο, ζουν στο Κουρδιστάν σε πάρα πολύ δύσκολε συνθήκες σε στρατόπεδα. Äh, και چادر και, που ακόμα ζουν στο βουνό ζουν σε πάρα πολύ κακές συνθήκες. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο να πάνε. I äh, Ελπίζω να θα μας βοηθήσετε ξαναχτίζοντας αυτά τα σχολεία. Η κυρία Μουράτ. Η κυρία Μουράτ. Η κυρία Μουράτ. Η κυρία Μουράτ. Η κυρία Μουράτ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για την ε, παρουσία σας εδώ, για το χρόνο που μας αφιερώνετε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που δεν ξέχασαν τι μας έκανε τον Ντάις και που μας υποστήριξαν. Πριν αρχίσω θα ήθελα να ευχαριστήσω το κρατήδιο τη Βάδης Βιρτεμβέργης που βοήθησαν τι ε, κοπέλε ε, από την κοινότητά μου και επέτρεψαν να κάνουν τη δουλειά που κάνω εγώ τώρα. Ελάχιστοι δεν γνωρίζουν τι είναι και τι κάνει το Ντάεσ. Γιατί δεν κρύβονται, είναι περήφανοι για τα εγκλήματα που κάνουν δημόσια, τα εγκλήματα ενάντια στις γυναίκες και τα παιδιά. دل روز و شب که دمالی از هەموو مبرین و نکب ابجیت مات مقدسێت کب دەها هاتی نەفەجراندن Για τρία χρόνια υποστήκαμε μεγάλες απώλειες, όχι μόνο υλικές, όχι μόνο τους ιερούς ναούς, α, αλλά ε, έγινε καταστροφή πνευματική. Σχεδόν όλες οι οικογένειες είχαν απώλειες μελών τους που είτε σκοτώθηκαν είτε υποδουλώθηκαν. Άρχισα το έργο μου αυτό πριν από ένα χρόνο. Από τότε που έφτασα στη Γερμανία, πρώτα ε, ε παρουσιάστηκα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να καταθέσω. Έχω επισκεφθεί 20 χώρες περίπου. Έχω συναντήσει πολλούς προέδρους, ε, βουλευτάς και άλλους αξιωματούχους.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 συνάντησα πάρα πολύ κόσμο. Τους κοίταξα κατάματα και τους μίλησα για τις χιλιάδες γυναίκες που πουλήθηκαν, που βιάστηκαν, που υποδουλώθηκαν, που έγιναν αντικείμενο ανταλλαγή. Μίλησα για όλα τα εγκλήματα της ISIS. Πολλές φορές ε, ντρέπομαι να επαναλαμβάνω τα ίδια.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

Θα πρέπει να υπάρξει λύση για όλες τις μειονότητες, μια ζώνη ασφαλείας και προστασίας που θα τις προστατεύει. Ε, οι, τις περιοχές των Γιαζίντι ε, θα πρέπει να τις προστατεύσουμε, αλλιώς ε, θα ε, διαφύγουν όλοι. Ε, Νομίζω ότι δεν πρέπει να ε, κατηγορηθούν όταν εγκαταλείψουν τη, τη, τα εδάφη τους ε, για να βρουν προστασία στην Ευρώπη. Δεν πρέπει κανείς να τις κατηγορήσει επειδή μεταναστεύουν.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

γιατί έδωσε ε, ευτυχία και περηφάνεια σε όλους μας στο Κουρδιστάν, στην Τουρκία, στην Ελλάδα έδωσε ευτυχία στην καρδιά όλων των θυμάτων σε όλο τον κόσμο. Πολύ ενθαρρυντικό αυτό και πολύ εγκαρδιωτικό ότι το βραβείο Ζαχάροφ ε, ανακουφίζει σε τόσο δύσκολους καιρούς ένα ολόκληρο λαό. Πριν λοιπόν ε, περάσουμε στη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο David Κάμπελ banderman που είναι ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Ιράκ. Θα μας πει λίγα λόγια για το, τι προσπάθειες κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση αυτή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και χαίρομαι ιδιαιτέρως που καλωσορίζω και εγώ μαζί σας τους δύο καλεσμένους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα θα έχουμε και μια επίσημη συνεδρίαση με την αντιπροσωπή για τη σχέση με το Ιράκ, παρουσία των καλεσμένων μας. Και εσείς στην Επιτροπή Εξωτερικών γνωρίζετε ότι το Ιράκ είναι το λίκνο του πολιτισμού. Βαβυλώνα είναι ακόμα εκεί και στη Βαγδάτη ε, ή τα ιστορικά μέρη της Συρίας και της Μεσοποταμίας και ε, και έχουμε Συρίους, ε, Τουρκμένους, Χριστιανούς και φυσικά έχουμε και τις κοινότητες Γιαζίντι που έχουν υποστεί τα πάνδυνα και ακούσαμε στην αντιπροσωπεία μας πολλές συνταρακτικές ιστορίες συνάντησα μία κυρία που είχε χάσει και τα τέσσερα της παιδιά από το Ισλαμικό κράτος και της φίλησα το χέρι γιατί ήταν το ελάχιστο που μπορούσα να κάνω απέναντι στην τεράστια θυσία που χρειάστηκε να κάνει. Οπότε αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό να καταστρέψουμε το αυτοποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος και ο Τσάρλς Τάνοκ ε, ε, επισκέφθηκε μαζί μου ε, την γραμμή των Πεσμεργά, 50 χιλιόμετρα από τη Μοσούλη και χαίρομαι που απελευθερώθηκε η Μοσούλη. Βέβαια ήταν πολύ δύσκολη η απελευθέρωση αυτή με σύραγγες, με βομβιστές αυτοκτονίας, με τρομοκρατικές επιθέσεις. Συγχαρητήρια για το βραβείο Ζαχάροφ, πραγματικά το αξίζεται. Και όπως είπα, θα κάνουμε μέσω τη αντιπροσωπεία μας πολύ περισσότερες προσπάθειες και θα έχουμε και την επίσημη συνεδρίαση αργότερα στην εβδομάδα μαζί σας. Ευχαριστώ θερμά για το έργο σα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές και μετά θα δώσουμε το λόγο και σε άλλους συναδέλφους. Από την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Κρύπ, για Τρία λεπτά κατά μέγιστον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τα πολωνικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τις γενναίες αυτές γυναίκες που εκπροσωπούν την κοινότητα των Γιαζίδη. Την κυρία Νάντια Μουράντ και την κυρία Λάμια Χατζιμπασάρ. Πραγματικά περάσατε από απίστευτα, αδιανόητα μαρτύρια. Μιλήστε ελάχιστα για τον εαυτό σας, μιλήστε περισσότερο για το λαό σας, για την κοινότητά σας. Και παρόλα αυτά τα μαρτύρια η ψυχή σας έμεινε αναλύωτη. Δεν σας έκαμψαν, γιατί το βραβείο Ζαχάροφ είναι το βραβείο της ελευθερίας σκέψης. Και γι' αυτό το ιδρύσαμε με τη συμφωνία του καθηγήτου Ζαχάροφ και νομίζω ότι αυτό το βραβείο σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει ε, τα μαρτύρια που έχουν υποστεί οι Γιαζιντοί ως κοινότητα. Αλλά όχι μόνο οι Γιαζιντοί και άλλες ε, θρησκευτικές μειονότητες που έχουν την επιτυχία να, να βρίσκονται στη ζώνη υπό τον έλεγχο του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους. Ήταν ε, τρομερές ε, οι διώξεις στο Γιαζίδι, των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων. Μερικοί χρειάστηκε να, να φύγουν για να γλιτώσουν, αναγκάστηκαν να, να αυτοεξοριστούν για να ξεφύγουν από τη δουλεία, τα μαρτύρια και το θάνατο. Και μάλιστα με πρωτοβουλία της ομάδας μας, στην αρχή του έτους, στα πλαίσια της συζήτησης των εγκλημάτων του ΝΤΑΕΣ, ε, χαρακτηρίσαμε αυτά τα εγκλήματα ως γενοκτονία και ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, και θα πρέπει να τιμωρηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γιατί υπάρχουν και αποδείξεις και τεκμήρια για τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και σας ευχαριστούμε θερμά για τη μαρτυρία σας, για αυτό που κάνετε προκειμένου να ε, γίνει παντού στον κόσμο ε, το, το μαρτύριό σας και αυτά που κάνουν στο Ισλαμικό κράτος. Έχουμε μαζί μας και άλλους φιναλίστ του βραβείου Ζαχάροφ. Τον, ε, είχαμε τον Τζαν Ντουντάρα, που έπρεπε να έρθει, αλλά έχουμε μαζί μας και τον Μουσταφά Τζεμίλεφ, που επίσης έφτασε στο τελικό στάδιο πριν την εκλογή και εκπροσωπεί του Τατάρους της Κρυμαίας και μάλιστα στις 2 Δεκεμβρίου, όταν έγινε μια συνεδρίαση παρουσία μου στη Βαρσοβία, μας είπε ο κύριος Τζεμίλεφ πολύ ωραία λόγια. Και όταν άκουσα ότι είναι και αυτός από τους φιναλίστ για το βραβείο Ζαχάροφ, σκέφτηκα πραγματικά αυτό είναι μια πολύ όμορφη αναγνώριση και σκέφτηκα ποια άλλοι θα μπορούσαν να είναι βραβευθέντες. Και είπα, ναι, αυτές οι δύο γυναίκες αναφυσβήτητα αξίζουν να λάβουν αυτό το βραβείο. Αυτό είπε ο, ο κύριος, ε, ο ίδιος ο Μουσταφά ε, Τζαμίλεφ. Νομίζω ότι και ο ίδιος αναγνώρισε πόσο σημαντικό είναι το έργο σας και πόσο άξιες είστε για την απονομή αυτού του βραβείου Ζαχάροφ. Και μάλιστα ο κύριος Τζαμιλεύ γνώριζε και προσωπικά τον καθηγητή Ζαχάροφ και μάλιστα ήταν τότε πολύ δύσκολη καιρή του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση και ο λαός του, οι τάταροι της Κρυμαίας υπέστησαν και τότε και εκείνη τα πάνδυνα από τη Σοβιετική Ένωση και τώρα έχουν πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να επιστρέψουν στις αιστείες τους, στην πατρίδα τους που ένα διάστημα είχαν επιστρέψει. Οπότε όλοι και οι δύο αυτοί φιναλίστ που αναφέρα ο κύριος Τζαντουντάρ από την Τουρκία και ο κύριος Τζεμίλεφ δεν βραβεύτηκαν με το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά πραγματικά βρέθηκαν ε, σε αυτή την ομάδα των εκλεκτών ανθρώπων που δίνουν μάχη για την ελευθερία σκέψης και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και σας ε, συγχαίρω θερμότατα και εσάς, αλλά και τους δύο άλλους φιναλίστ στο βραβείο Ζαχάροφ. Σας ευχαριστώ θερμά. Um, Εμείς ευχαριστούμε για τώρα το λόγο του κ. Παντζέρη για τη σοσιαλιστική ομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να πω από πλευρά σοσιαλδημοκρατών ότι αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνεια διότι σήμερα έχουμε εδώ την Άντια Μουράτ και την κυρία Λαμία Χατζιμπασάρ. Βρίσκονται εδώ για να τους απονείμουμε το βραβείο Ζαχαρόφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πέραν του καλωσόρισαν επίσης και οι δύο φινελίστες, ο κύριος Ντουντάρ και ο κύριος Τζεμίλεφ, θα πρέπει να ξέρουν ότι θα έχουν την αμέριστη υποστήριξή μας. Η Νάντια και η Λάμια έχετε περάσει τις πιο φρικτές εμπειρίες. Κάτι που δεν πρέπει να περνά κανείς άνθρωπος στη διάρκεια της ζωής του. Όλοι σε αυτή την αίθουσα θαυμάζουμε το πώς αντιδράσατε με τέτοιο ευγενή τρόπο ευγενή από πλευράς ηθικής. Από θύματα γίνατε μαχητές, μαχητές κατά των εγκλημάτων του Ισλαμικού κράτους με αυτή την θεολογία της βίας το, που υφίστανται οι ανήλικοι και οι γυναίκες των Γεζίδη. Πρόκειται για κρίματα, για, συγγνώμη, για εγκλήματα τον Αύγουστο του 2014 στα χωριά σας, κοντά στο σύνομα τη Συρία, στο βορειοδυτικό Ιράκ. Και τον Ιούνιο του 2016 Αποκαλύφθηκε και αυτό το ε, έγκλημα, αυτή η γενοκτονία κατά τον Γεζίντη, που είναι ένα έγκλημα πολέμου, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά των ανηλίκων, κατά των ε, γυναικών που με τη βία συρρόντουσαν στο Ιράκ και στην Συρία. Και εκεί είναι ακόμα φυλακισμένοι. Επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε αυτή την συστηματική χρήση του βιασμού ως όπλο πολέμου και έχει ελκύσει την προσοχή σε αυτές τις φρικαλίωτες που δεν είναι μόνο εγκλήματα πολέμου, είναι μέρος μιας στρατηγικής. Οπότε θα πρέπει όλα αυτά να τιμωρούνται ως εγκλήματα πολέμου. Και το 2014 είχαμε τον Δόκτωρα Μουγγέβε που αναδείξαμε το έργο του για τα όσα έκανε στο Κονγκό. Οπότε θα πρέπει, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, να βοηθήσουμε να μην υπάρχει πια ατιμορρησία για όσους διέπραξαν τέτοια εγκλήματα, για όσους απειλούν την ε, ασφάλεια, για όσους κάνουν αυτά τα ε, εγκλήματα πολέμου και όλοι αυτοί θα πρέπει να συρθούν ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σήμερα μας ε, είπατε για το πώς μπορούμε να συσπηρωθούμε, πώς είναι δυνατόν ε, να προχωρήσουμε και την ε, Πέμπτη επίσης θα έχουμε ένα ψήφισμα για τους κοινού ε, τάφους του Ιράκ. Αγαπητές βραβευθήσεις με το βραβείο Ζαχάρου θα πρέπει για άλλη μια φορά η πολιτική μας ομάδα να σας ε, συγχαρεί. Θα πρέπει να σας πούμε ότι έτσι θα γίνετε πιο δυνατές. Έτσι ο ρόλος σας θα προβληθεί περισσότερο, θα αποκτήσει περισσότερη σημασία. Θα εκφράσετε και θα κάνετε να ακουστεί η φωνή των ζήτη, κυρίως των γυναικών. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω θερμά κυρία Πρόεδρε τις ε, καλεσμένες μας απόψε εξ ονόματος της ομάδας ECR, την τρίτη ομάδα του Κοινοβουλίου, τις κυρίες Μουράντ και Χατζή Μπασάρ Χαιρετίζω θερμά ε, και τον κύριο Τζεμίλεφ που τον γνωρίζω εδώ και καιρό και είχα την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω όταν ήρθε στην ομάδα μας ε, στις Βρυξέλλες ε, και τον ευχαρίστησα για ό,τι κάνει για τους Τατάρους στην Κρυμαία. Θέλω να καλωσορίσω τις προσκεκλημένες μας για Ζήντη και να τις συγχαρώ για το βραβείο Ζαχάροφ 2016. Είχα την ευκαιρία, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος David Campbell Bannerman πριν από λίγο, να ε, επισκεφθώ το Ιρακινό Κουρδιστάν και χάρηκα διότι υποστήριξα αίτημα που απευθύνθηκε σε μένα όταν ήμουν επικεφαλής από τον πρόεδρο Μπαρζάνη από την KIG και πιστεύω και κατάλαβα ότι οι Γιαζίδοι θεωρούν τον εαυτό τους ε, ως αρχαίο κουρδικό πολιτισμό ε, δηλαδή ε, είναι κοντά στους Κούρδους. Ο κύριος ε, μου ζήτησε να ασκήσω πιέσεις στις κυβερνήσεις, κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας, να θέσω το θέμα στον Βρετανό πρέσβη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ούτως ώστε να παρα πενθεί στο Διεθνές Δικαστήριο ο ΑΕΣΙΣ ε, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Του ε, υπεύθυνου ε, τους υπεύθυνους ε, για τη γενοκτονία την απόπειρα γενοκτονίας κατά τον Γιαζίντη. Δεν με υποστήριξαν πολύ για λόγους που δεν είναι απόλυτα σαφείς. Ελπίζω το βραβείο Ζαχαρόφ να αλλάξει πολλές απόψεις στα, ε, στους Γάλλους και Άγγλους ε, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, ως υπεύθυνο για τις για το Κουρδιστάν είχα υποδεχθεί ε, πολλούς γιαζίδεις σε συναντήσεις και υπήρχαν και, ήρθαν και μαχητές πεσμεργά που όπως οι κυρίες σήμερα πέρασαν πολλά δεινά στα χέρια των μαχητών του ISIS και ε, εντυπωσιάστηκα από το θάρρος των Γιαζίδη που ε, υπέστησαν τα πάνδυνα ε, από τον Άισις ε, υποδούλωση των γυναικών, μαζικές εκτελέσεις ε, των ανδρών μελών οικογενειών μπροστά στις γυναίκες και τις, τα παιδιά τους. Ήταν ε, μία από τις μεγαλύτερες ομότητες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή. Και οι δύο βραβευθύσες υπέστησαν πολλά στα χέρια του των υπεύθυνων του και πιστεύω ότι θα ε, αποτελέσουν σύμβολο που θα εμψυχώσει την κοινότητα των Γιαζίντι και θα συνεχίσουν να βοηθούν με τον τρόπο αυτό τις γυναίκες και τα παιδιά που παραμένουν σε εχμαλωσία και υποδούλωση από τον Άισις και τώρα που μιλάμε στην Ράκα, στη Μοσούλη και σε άλλα ελεγχόμενα εδάφη ε, υπόκεινται σε τρομερές ομότητες. Ελπίζομαι ότι σύντομα θα δούμε το τέλος του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους ε, η Διεθνής Συμμαχία ε, κλιμακώνει τις πιέσεις και ελπίζω ότι ο ISIS Daesh θα καταστραφεί και θα εξαλειφθεί από την περιοχή το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ οι συνάδελφοι συμφωνούν με τις ε, τελευταίες παρατηρήσεις σας. Η Μπεατρής Μπεσέρα από τους Φιλελεύθερους. Σας ευχαριστώ. Αγαπημένες μου Νάντια και λάμια. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μπορεί να μην το πρόφερα σωστά, αλλά ήθελα να το πω. Συγχαρητήρια. Τα καταφέραμε. Ήταν μακρύς ο δρόμος μέχρι να φτάσουμε εδώ, αλλά είστε μπροστά μας ε, οι βραβευθύσεις που μας φωτίζετε ως φάρι. Θυμάμαι την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, Νάντια, το Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες και πραγματικά με συντάραξε, με συγκλώνησε η ιστορία σου και η αποφασιστικότητά σου και ανέλαβε απέναντί σου μία δέσμευση και μία ευθύνη. Αργότερα γνώρισα και τη Λάμια στο Στρασβούργο μέσω του συναδέλφου μου του κ. Βάιντεν Χόλτσερ και οι μαρτυρίες σας με ενέπνευσαν για το έργο μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ θερμά. Και από τη μέρα που σε γνώρισα, Νάντια, κατάλαβα ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσω κάθε μέσο ότι είχα στη διάθεσή μου για να σε βοηθήσω, να σε βοηθήσω στον αγώνα σου. Και γι' αυτό ακριβώ ε, αποφάσισα να καταθέσω την υποψηφιότητά σου για το βραβείο Ζαχάροφ. Γιατί είναι ένα μοναδικό, καταπληκτικό, εξαιρετικό εργαλείο, ένα μέσο για να μάθει ολόκληρο ο κόσμο την ιστορία σα για ε, να σας δώσει και μια οικονομική ενίσχυση για να υλοποιήσετε το στόχο σας, ε, που είναι το όραμά σας, να φέρετε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τη γενοκτονία που διαπράττει το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος εις βάρος του λαού σας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί μπροστά σας βλέπω να αντικατοπτρίσετε η υπέρβαση, η ιστορία της υπέρβασης της ευρωπαϊκής ιστορίας, που ξεπέρασε τρομερές θηριωδίες και βαναυσότητες, απερίγραπτες και απίστευτες. Μόνο ένας άνθρωπος με ξεχωριστή δύναμη μπορεί να τις ξεπεράσει χρησιμοποιήσατε πάντω την οδύνη σα για να κάνετε κάτι που ξεπερνάει εσάς τι ίδιε και να προστατεύσετε τα στοιχειώδη δικαιώματα του λαού σα και να καταγγείλετε το γενο, τη γενοκτονία στις, ε, στα ύψιστα κλιμάκια και στη, στα ισονότερους βαθμού τη δικαιοσύνη. προκειμένου να βρείτε τελικά την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Νάντια και Λαμία, χτίστηκε στις τάχτες τη βαρβαρότητας ε, ανάμεσα σε λαούς που ενώ βρίσκονταν μεταξύ τους σε σύραξη τελικά αποφάσισαν να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους τα δικά τους οράματα και να κοιτάξουν πιο μακριά. Και μάλιστα ο Μέγας Βίκτορ Ουγκό το είπε πολύ σωστά. Θα έρθει μια μέρα που οι βόμβες θα αντικατασταθούν από την αξιοσέβαστη διατησία κυρία τη Γερουσία που θα γίνει και την Ευρώπη ό,τι είναι η Εθνοσυνέλευση και τη Γαλλία. Το βραβείο Ζαχάροφ αποτελεί την ψυχή του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου και την ενσάρκωση των αξιών και αρχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την ελευθερία, την ε, δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος ε, δικαίου, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εσείς, Νάντια και Λάμια, εκπροσωπείτε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο τις αξίες για τις οποίες αγωνιζόμαστε στην Ευρώπη. Και γι' αυτό αξίζεται αυτό το βραβείο. Και επαναλαμβάνω και διατρανώνω την δέσμευσή μου απέναντί σας και απέναντι στο λαό για ζητή. Γιατί τώρα αρχίζει ο δρόμος μας. Πάνω από 3.000 γυναίκες και κορίτσια εξακολουθούν να είναι υποδολουμένες και να βιώνουν καθημερινά το γολγοθά που ζήσετε κι εσείς. Γνωρίζεις μπορεί, ότι μπορείς να υπολογίζεις ε, στην, ε, στην δεσμευσή μου, την αμετάκλητη, για να σου συμπαρασταθώ σε αυτή την επίμονη προσπάθειά σου να φέρει τον ΤΑΕΣ μπροστά στο Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Και ω Αντιπρόεδρο τη Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω εκ βάθου καρδία για τον αγώνα σα. Σα ευχαριστώ που είστε παράδειγμα προ για τον κόσμο όλο, γιατί και εμεί, η Ευρώπη, ο κόσμο, χρειαζόμαστε περισσότερε συνάντειε, περισσότερε λάμιε, περισσότερου Ζαχάρο. Σα ευχαριστώ. Κύριε Μακάβαν, σας ευχαριστούμε εμείς και τώρα έχει το λόγο η κυρία Βερζιάτ για την Γκουε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μπαίνει μου χαρά σας λέω εδώ. Αυτή τη βδομάδα που ήρθατε για να σας απονεμηθεί το βραβείο Ζαχάροφ και εγώ όπως και οι άλλοι Συμπαθάτε με λέει Αλλά τέλο πάντων θέλω και εγώ να ενώσω τη φωνή μου. Τόσο άλλοι για αυτή την ε, εβδομάδα που είχαμε τον κύριο Ντουντάρα αλλά και τον ε, κύριο Τσέντιν διότι νομίζω ότι αυτοί που ήταν οι φιναλίστ και αυτοί άξιζαν το βραβείο Ζαχάροφ. Αυτά τα οποία πάθατε τα πάθατε για τους εξής τρεις λόγους ως γυναίκες. Δεύτερον, λόγω της ε, θρησκείας σας και τρίτον γιατί πάρα πολλοί από τους Γεζίντε είναι Κούρδοι. Να μην είπαν αυτά που είπαν ε, οι άλλοι για αυτές τις φρικαλότητες που υπέστητε γιατί μόνο που τα λέει κανείς είναι σαν σας μαχαιρώνει στην καρδιά, δεν αξίζει. Ναι, πρόκειται για γενοκτονία, πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα κατά της γυναίκας, εγκλήματα πολέμου. Και εγώ εκπροσωπώ εδώ την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και θέλουμε να χαιρετήσουμε το θάρρος σας. Για το ότι τώρα δίνεται αγώνα για να αναγνωριστούν αυτά που έγιναν στο παρελθόν και για να απελευθερωθούν εκείνοι που είναι ακόμα στα χέρια των ε, βαρβάρων, για τον αγώνα που δίνεται για την ειρήνη. Γιατί νομίζω ότι σε εκείνη την περιοχή του κόσμου αυτό το οποίο χρειάζεται είναι όσο περισσότεροι να δίνουν μάχη για την επικράτηση της ε, ειρήνης πάνω από κάθε χειραγώγηση που τόσο συχνά συμβαίνει σήμερα. Οπότε ε, ευχαριστούμε και πάλι ευχαριστούμε και πάλι μπράβο για το θάρρος σας. Είσαστε παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα των Πρασίνων. κυρία, οι κυρίες Λόχμπιλερ και Χάουταλα θα μοιραστούν το τρίλεπτο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Καλώς ήρθατε και ένα θερμό ευχαριστώ κυρίες ε, Μουρατ και Χατζιμπασάρα. Παρόλα τα δεινά που υποστήκατε, προχωρήσατε, παρουσιαστήκατε μπροστά στην κοινή γνώμη και δίνετε μάχη για την απελευθέρωση και των άλλων γυναικών. Η κυρία Χατζή Μπασάρα αναφέρθηκε σε μια απόφαση του Φεβρουαρίου φέτος του Κοινοβουλίου, όπου ασχοληθήκαμε με την κατάσταση στο Ιράκ και στο ψήφισμα είχαμε ζητήσει, μεταξύ άλλων, ότι αν υπάρξει πολιτική ε, δίκη για την περιοχή θα πρέπει θα πρέπει να αρχίσει μια πολιτική διαδικασία στην περιοχή, ούτω ώστε να ε, επιτευχθεί μια σταθερή, μια διαρκή λύση. Ελπίζω και εσείς να, μετέχετε στη διαδικασία αυτή. Είπατε κυρία Μουράτε ότι είναι σημαντικό να ταυτοποιηθούν, να αναγνωριστούν και να λογοδοτήσουν οι υπέτειοι. Αυτή τη βδομάδα σε ένα ψήφισμά μας ζητούμε ε, η μαζική ε, τάφη ε, να, στο, στην περιοχή Σιντζάρ να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Το Κοινοβούλιο έδωσε, δίνει μάχη γι' αυτό και τώρα θα πρέπει να απευθυνθεί έκκληση στον Πρόεδρο ούτως ώστε να προσπαθήσει και εκείνος. Ε, δέχομαι την ευχαριστία σας προς το κρατήριο Βάδη Βιρτεμβέργη. 600 ε, γυναίκες βρίσκονται εκεί, στο κρατήριο αυτό και υπάρχει ε, υποστήριξη ε, και από το Πανεπιστήμιο για την αντιμετώπιση του μετατραυματικού στρες εκτός από την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Ε, η βοήθειά μας πρέπει να είναι γενναιόδορη ε, στον τομέα της ιατρικής και της ψυχολογίας, της βοήθειας που πρέπει να δοθεί και θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη όσο τα δεινά που υποστήκατε. Και εγώ ε, θα ήθελα, κυρία Πρόεδρε, να, να καλωσορίσω τις κυρίες Νάντια Μουράτ και Λάμια Χατζιμπασάρ στο Κοινοβούλιο. Ε, όταν η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Νομική Επιτροπή συζήτησε διάφορες εναλλακτικές για το πώς η ε, στιγμή αυτή εγκληματίες της ΤΑΕΣ να προσέλθουν στο δικαστήριο και μία εναλλακτική που συζητήθηκε ήταν να δούμε μήπως θα έπρεπε να υπάρξει ε, έξω εδαφικότητα. Κάποια κράτη-μέλη ε, ε, εντόπισαν ως ε, μαχητές της ΔΑΕΣ που είχαν επιστρέψει και ίσως η ετεροδικία θα πρέπει να είναι η βραχυπρόθεσμη λύση ούτως ώστε να λογοδοτήσουν οι υπέτοιοι. 104 μέλη του Κοινοβουλίου ήδη τον Απρίλιο απίφθηναν στην κυρία Μογκερίνη επιστολή ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ε, να ε, αναδείξει ε, το πρόβλημα ως γενοκτονία. Ήδη είχαμε διατυπώσει έτοιμα στην κυρία Μογκερίνη από το Σεπτέμβριο, αλλά δεν είχαμε απαντήσει. Ίσως αυτή τη βδομάδα η κυρία Μογκερίνη να απαντήσει σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, γιατί πρέπει να φροντίσουμε να προσαχθούν στην δικαιοσύνη οι υπέτειοι. Ε, και ε, αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό όταν αποδειχθεί η γενοκτονία. Ο Φάμπιο Καστάλντο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, και εγώ δεν μπορώ παρά να συμμεριστώ τα όσα είπαν οι συνάδελφοι για την ε, Νάντια και την Λαμία. Για το ήρθαν εδώ να μας καταθέσουν τον αγώνα τους και να πω το πόσο επίσης ε, θαυμάζουμε τον ε, Ντούνταρ και τον ε, Τζέμιλαφ, τους υποψηφίου που δεν μπορούσαν να είναι και εδώ και οι δύο για να μας πούνε τι γίνεται ο κύριος Ντουντάρ δηλαδή για την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία σε αυτές τις δύσκολες ώρες της σχέσης μας με τη χώρα εκείνη. Μα είπατε επομένω και οι δυο σα τι γίνεται με του βιασμού, με τη σεξουαλική δουλεία όλα αυτά τα οποία ναι τα, ξέρουμε αλλά υπάρχουν και χειρότερα πράγματα εκεί αυτή η φτώχεια του ότι δεν υπάρχουν ε, που ε, δεν υπάρχουν που σπανίζουν στην διεθνή κοινότητα που είναι η σιωπή και η αδιαφορία άλλες είναι πατριώτες της κοινότητας οπότε ε, τόσο καιρό το δράμα των Γεζιτή είναι κάτι που το ζουν μόνο οι ίδιοι οι Δεν έχει γίνει όσο γνωστό θα έπρεπε, γιατί υπολογίζονται πάνω από 3.000 οι ανήλικοι και οι γυναίκες που είναι φυλακισμένοι από το Ισλαμικό κράτος. Πάρα πολλοί έχουν αυτοκτονήσει. Γονάτισαν οι οικογένειες για λόγους οικονομικούς, οπότε πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Όχι δεν μπορούμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κάνουμε όμως ένα μικρό πρώτο βήμα να απονείμουμε αυτό το βραβείο. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να αντιδράσουμε όπως επιβάλλεται είναι το να απονείμουμε δικαιοσύνη. Έχουμε κατεπήγον ψήφισμα να εγκρίνουμε όσον αφορά αυτούς τους κοινού τάφους. Θα πρέπει όμως οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα να προσταθούν στη δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να κάνει η διεθνή κοινότητα. Και επίσης θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί η πατρίδα σα και να αντιμετωπιστεί το θέμα του κινδύνου τη επιστροφή. Το σκεφτόμαστε και ξέρουμε ποιε είναι οι συνθήκε εκεί. Το πιο σημαντικό, επομένως για σας, είναι να υπάρξει ξανά εκεί η ελευθερία, η ομαλότητα και το χαμόγελο στα χείλη των παιδιών. Αυτό πρέπει να κάνει το Κοινοβούλιο πιέζοντας τις κυβερνήσεις. Γιατί αν δεν υπάρξει αποφασιστική δράση και θέληση δεν θα υπάρξει ούτε ειρήνη, ούτε δικαιοσύνη. Ούτε για τη Συρία, ούτε πουθενά άλλο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε και όλα τα άλλα θύματα. Ευχαριστούμε που τώρα τους δίνετε την ευκαιρία να περπατούν με το κεφάλι ψηλά θύματα αυτών όλων των βαρβάρων που το κάνουν χωρίς καμία δικαιολογία. Σας ευχαριστούμε κύριε Καστάλτο. Και τώρα ο κύριος Λορέντσιου Ρεμπεγκά από την ομάδα ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλεσμένοι. Ε, είναι υποδειγματική η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απονομή του βραβείου Ζαχάροφ δεν είναι μια απλή τελετουργία, αλλά αυτή η απόδειξη της δέσμευσης των Ευρωβουλευτών απέναντι στις οικουμενικές αξίες ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, αποφασίσαμε να απονείμουμε φέτος ε, το βραβείο Ζαχάροφ 2016 στην Άντια Μουράτ και στην Λάμια Μπασάρ που δυστυχώς δείχνουν το πιο σκοτεινό πρόσωπο της σημερινής πραγματικότητας του εμπορίου ανθρώπων και της σεξουαλικής δουλείας. Μέχρι στιγμής ε, η παγκόσμια κοινότητα φαίνεται ότι αγνοούσε η ε, θελοτυφλούσε προς τα, πράγματα, προς τα φαινόμενα. Εμεί δείξαμε ότι θα πρέπει να πρετανεύσει η ανθρωπιά και να, ε, να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα του 21ου αιώνα που είναι η τρομοκρατία μαζί με, την, με τις συμπαρομαρτούσες βαναυσότητες και τις θηριωδίες της γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από έναν θρησκευτικό φανατισμό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για τη θρησκεία εδώ. Και το πρόβλημα σήμερα δεν είναι μεταξύ των θρησκειών. Είναι η αντιπαράθεση των θρησκειών και του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα, στη βαναυσότητα. Γιατί είναι όλα μία πάλι για την ανάκτηση εξουσίας. Και δυστυχώς τα θύματα πάντα είναι οι ειρηνικοί, φιλοιρηνικοί άνθρωποι, άμαχος πληθυσμός, οι καλοί άνθρωποι. Και η Νάντια Μουράτ και η Λάμια βασάρ είναι τα σύμβολα αυτής της μάχης υπέρ του ανθρωπισμού και είναι ηρωίδες απέναντι στα μαρτύρια που πέρασαν και δίπλα τους υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλες γυναίκες που σε διάφορα μέρη του κόσμου επίσης είναι θύματα της σεξουαλικής υποδούλωσης και της σωματεβορίας. Και τα σημερινά γεγονότα θα πρέπει να μας αφυπνήσουν ώστε να αναλάβουμε δράση και να εξαλείψουμε αυτή τη μάστιγα. Θα πρέπει να αφήσουμε ένα καλύτερο κόσμο στις επερχόμενες γενιές. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το κακό με την αδιαφορία ε, γιατί το κακό εδράζεται στον πόλεμο, στην κατάργηση των αξιών, στην δημιουργία φόβου και μίσους γιατί ε, μόνο το δίκαιο του δυνατού επικρατεί στον πόλεμο. Και δεν χρειάζεται μεγάλη οξυδέρκεια για να δούμε ότι τέτοιου είδους σωματεμπορία και σεξουαλική υποδούλωση ανθεί κυρίω σε εμπόλεμες ε, περιοχές, ε, σε ζώνες που βρίσκονται στη σειράξη. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας γιατί από την απεικιοκρατική εποχή είχαμε τέτοια φαινόμενα και άλλες φορές τα οικονομικά συμφέροντα ή γεωπολιτικοί ε, κοινικοί λόγοι προκάλεσαν άνθηση τέτοιων φαινομένων. Θα πρέπει να πατάξουμε επιτέλου να σταματήσουμε αυτά τα φαινόμενα και να δράσουμε το συντομότερο δυνατό για να σταματήσουμε τον πόλεμο και να εξαρθρώσουμε την τρομοκρατία. Δεν είναι φυσικά κάτι τέτοιο εύκολο, αλλά είναι ο μόνος δρόμος. Και μάλιστα σε συντρίμια ε, των ε, πόλων αυτών είναι φυσικό να ε, αλληλοσκοτώνονται όσοι απομένουν εκεί για να επιβιώσουν. Θα πρέπει λοιπόν στα συντρίμια αυτά να φτιάξουμε υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία, ε, να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν, να βρουν μια δουλειά και να αρχίσουν να εκτιμούν ο ένας τον άλλο και να συνεπάρχουν ειρηνικά. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει λύσεις ειρήνης, ε, ευμάρειας και πολιτισμού. Χαιρόμαστε για την απονομή αυτού του βραβείου Ζαχάροφ ε, για αυτές, σε αυτές τις δύο γυναίκες που είναι σύμβολα αυτού του αγώνα ώστε να αποτραπεί ε, η γενίκευση αυτών των φαινομένων. Uh, Πέντε άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, αλλά παρακαλώ να είστε λακωνικοί, γιατί θέλω να μείνει χρόνος να ακούσουμε τον κύριο Τζεμίλεφ. Η κυρία Χιμένες Μπεσερίλ και μετά ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάθε απονομή του Βορείου Ζαχαροφ είναι απονομή προς κάποιον ο οποίος το αξίζει, αλλά και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ε, το, αξίζουν 500% και ακούσατε τι είπανε, είναι πάρα πολύ ε, Έχουμε αυτή την ταπείνωση από το Ισλαμικό κράτος, έχουμε τους διασμούς από το Ισλαμικό κράτος, οπότε πάρα πολύ συγκινήθηκα σήμερα μας ευχαριστήσατε που ήρθαμε εδώ, που ε, αναλώσαμε το χρόνο μας. Μα εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό μέρος να βρίσκεται κανείς σήμερα από το να βρίσκεται εδώ για να σας ευχαριστήσει για όλα όσα κάνατε. Ε, κοιτάξτε, ε, από κάθε τραγωδία κάτι βγαίνει και είναι αυτό το, τώρα, αυτό το κίνητρο που μας δίνεται ε, δηλαδή το, η θέληση της ζωής κάτι να κάνουμε για τα θύματα, να δείξουμε στους τρομοκράτες ότι κάνανε ε, πάρα πολύ μεγάλο κακό, αλλά δεν μπορούν να κάνουν παραπάνω. Και αυτό το δείχνετε εσείς που είσαστε εδώ σήμερα και η διαφορά, ε, η διαφορά μεταξύ οδήποτε εγκλήματος και της τρομοκρατίας είναι ότι οι μόνοι εγκληματίε οι οποίοι νιώθουν περήφανοι και δημοσιοποιούν τα όσα κάνουν είναι οι τρομοκράτε. Άρα και εμεί ακριβώ να κάνουμε να ακουστεί η φωνή των θυμάτων και να ακούγεται λιγότερο η φωνή των τρομοκράτων. Και να κατακλείδη να σα πω δεν είσαστε μόνε. Το Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια προσπαθεί με, με, με ψηφίσμα να υποστηρίξει τι ε, ε, χριστιανικέ μειοψηφίε όπω Και ε, ε, όπως όπω ακούσατε έχουμε και αυτό το ψήφισμα για τους γενοστάφους. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατευτείτε, να γυρίσετε ε, στην πατρίδα σας και θα πρέπει να προστατεύουμε τα δικαιώματα των θυμάτων παντού και στο Ιράκ, παντού όπου χτυπάει η τρομοκρατία. Το δικαίωμα στην ε, ελευθερία, στη δικαιοσύνη, στην ε, μνήμη και στην αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς, λέει κυρία Μακάβων. Και τώρα ο κύριος Χόλτσερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ομάδας φιλίας ε, με τους Γιαζίντις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δύο βραδευθύσεις. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, εδώ στο Κοινοβούλιο για την υποστήριξη. Ελπίζω να συνεχιστεί και να είναι πολυάριθμη. Θυμάμαι ακριβώς τη μέρα, εδώ στην αίθουσα αυτή ακριβώς, όπου εξ ονόματος της ομάδας μου μπόρεσα να παρουσιάσω την σχετική πρόταση. Και όταν τελείωσα την παρουσίαση μου, ε, πήρα ένα SMS και έμαθα ότι είχα γίνει παππούς ενός μικρού αγοριού. Ε, συγκινήθηκα όταν σκέφτηκα πόσο η χαρά και ο πόνος είναι ε, αλληλένδετα και νομίζω ότι ήταν και παράλληλα ένα καλό μήνυμα, ένα προ... μήνυμα ότι ε, θα συμβεί κάτι καλό, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Τον Αύγουστο του 2014 ε, ε, άρχισαν οι διώξεις, οι γενοκτονίες, ε, ένας αριθμός κλιμακούμενων ε, συμφορών και νομίζω ότι θα πρέπει αποφασιστικά να αντιδράσουμε. Το σκέφτομαι καθημερινά αυτό. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση ιερή να βοηθήσουμε τον κόσμο αυτό να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Ε, δεν ξέρω αν θέλουμε να μιλήσουμε για αυτοδιοίκηση, για αυτοδιάθεση. Οι μειονότητε όμως θα πρέπει να έχουν μια ανεξαρτησία μαζί με τους χριστιανούς ε, φίλους με τους οποίους ε, συμβίωσαν τόσο αρμονικά επί ε, χρόνια. Ε, πριν από τρει εβδομάδε ε, πήγα στην Ελλάδα και είδα ε, που ε, μέχρι πρόσφατα ζούσαν σε σκηνές, σε καταβλισμούς, ε, στο χιόνι ε, πριν από λίγο καιρό μετά από όλες αυτές τις διώξεις και στην Ευρώπη όπου έφτασαν πολλοί και βρήκαν προστασία και στην κάτω Σαξονία αρκετοί από αυτούς και βλέπω ότι όλοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν βοήθεια ε, στους συμπατριώτες τους. Ε, χαίρομαι για αυτή την ε, αερογέφυρα που δημιουργήθηκε για να φτάσουν στην Γερμανία και να απολαύσουν κάποια δικαιώματα. Θερμή παράκληση να ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη το παράδειγμα της ε, Βάδης Βιρτεμβέργης. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και θα πρέπει να υπάρχει και συμφιλίωση. Ε, μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό σήμερα, αλλά αν δεν υπάρξει και συμφιλίωση ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτε. Ε, η Λάμια όταν συναντηθήκαμε μου διηγήθηκε την απαγωγή της. Πριν την απαγωγή θέλει να γίνει ε, δασκάλα. Ελπίζω να τα καταφέρει και ελπίζω ε, όλες οι γυναίκες για ζήτη ε, να γίνουν ε, εκπαιδεύτριες σε θέματα ανθρωπισμού και συμπόνιας. Ευχαριστώ. Σας έδωσα περισσότερο χρόνο, διότι εσείς κάνατε την πρόταση ε, για το βραβείο Ζαχάροφ. Ε, έχουμε δύο λαμπερά παραδείγματα για ζήτη ε, που ε, βοηθήθηκαν από την υποστήριξη τη δική μας. Κύριος Αντάκτουσον, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τις διαβραβευθήσεις με το βραβείο Ζαχάροφ. Να σας καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να σας ευχαριστήσω που μας διηγηθήκατε την ιστορία σας με τέτοια γενναιότητα και με τόση αξιοπρέπεια, ώστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι τις αποτρόπες ε, εμπειρίες που βιώσατε. Είχα το προνόμιο να είμαι από τους αρχικούς συντάκτες ε, αυτού του ψηφίσματος του Φεβρουαρίου που μίλησε για τις ε, βαναυσότητες, τις θηριωδίες και τις διώξεις ε, κατά των ε, γεζίδι χριστιανών και το χαρακτηρισμό τους ως γενοκτονία. Ήταν ιστορικό αυτό το ψήφισμα γιατί πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε μία γενοκτονία όσο γίνεται και μετά την αναγνώριση αυτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησαν και άλλες εθνικές βουλές. Για παράδειγμα, η Βουλή των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας ή η βουλη των Αντιπροσώπων και η Γερουσία στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και ο Λευκός Ήχκος ακολούθησε, μας μιμήθηκε και αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πραγματικά λοιπόν είναι σπουδαία αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η στιγμή και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανο γιατί κάθε φορά που πήγα στο Ιράκ, τρει φορέ πήγα στο Ιράκ του τελευταίου 15 μήνε και διαπιστώνω με χαρά ότι όλοι γνώριζαν το ψήφισμα αυτό που υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σημαίνει πολλά αυτό το ψήφισμα για τα θύματα αυτή τη γενοκτονία. Αυτή η αναγνώριση σημαίνει πολλά. Και φυσικά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και να φροντίσουμε ώστε όλα όσα και άλλες χριστιανικές μειονότητες και άλλες ομάδες να μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους αιστείες και στις πατρίδες τους. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της και να διευκολύνει την επιστροφή αυτή και να την καταστήσει δυνατή. Και χαίρομαι γιατί συγκεντρώσαμε μεγάλη διακομματική πλειοψηφία υπέρ της υποστήριξης μιας αυτόνομης περιοχής που θα πρέπει να επικεντρωθεί στην περιοχή Σιντζάρ και στην περιοχή Ταλαφάρ, στο Ιράκ. Θα πρέπει λοιπόν με αυτή την πρωτοβουλία να συνεχίσουμε και σας διαβεβαιώ ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, θα συνεχίσουμε μέχρι ότου πραγματοθεί αυτή η επιθυμία σας και επιστρέψετε στις αιστείες σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι που ήρθατε και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Σας ευχαριστούμε κύριε Δάκτουσον. Η Γκόμες. Λαμία, ε, σε ευχαριστούμε και σένα, Νάντια. Ευχαριστούμε τον κύριο Τζεμίλεφ και τον κύριο Ντοντάρη και είναι εδώ. Μια που έλαμψαν, δίνοντα αυτό το παράδειγμα για τον αγώνα που έδωσαν και που δεν κατέδεσαν τα όπλα. Ότι ευχαρίστησε η Νάντια το κρατήριο της Βάδης ε, Βιτεμβέργη για το πρόγραμμα αυτό ε, που βοήθησε την σωτηρία γυναικών και παιδιών και που τους ε, επέτρεψε να περάσουν από κάποια θεραπευτική διαδικασία. Γιατί το έκανε αυτό το κρατήριο της Βάδης Βιτεμβέργη και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Μαρία Σχάγε την την Κονελία Έρνστε που είχαμε πάει στο Βορειο τον Ιανουάριο του 2015 και αυτά τα αναφέραμε. Απευθυνθήκαμε στον εκπρόσωπο τη κυρία Μαγκερίνη ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία για να σώσει τι γυναίκε αλλά και τα παιδιά που βρισκόντουσαν στα χέρια των τζιχαντιστών και να υπάρξει βοήθεια, να υπάρξει θεραπεία για αυτά τα τραύματα που υπέστησαν. Γιατί δεν αναβάλει μια άλλη πρωτοβουλία πέραν της στρατηγικής βοήθειας από τους μερικά; Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, αναλαμβάνει πρωτοβουλία συντονιστική και να εξασφαλίσει ότι το Σιντζάρ τώρα θα ξαναχτιστεί και θα έχει την απαραίτητη ασφάλεια του ώστε κόσμο να ξαναγυρίσει στον τόπο του. Μα γιατί να μην ακούγεται περισσότερη φωνή τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη δικαιοσύνη, το διεθνέ ποινικό δικαστήριο, τι εισαγγελικέ αρχέ, τι διοικητικέ αρχέ τέλο πάντων. Γιατί αφού διαπιστώνουμε και ξαναδιαπιστώνουμε ότι είναι γεγονός το το εγκληματή τη γενοκτονία κατά τον Γιαζίδη. Γιατί να μην υπάρχει όλη αυτή η δυσμενή διάκριση ει βάρο των Γιαζίδη. Το είδαμε αυτό στου καταβλισμού των προσφύγων στην Ελλάδα με τον Ιώζεφ. Όλε αυτέ οι ερωτήσει απευθύνονται σε εμά, του εαυτού μα, να το αναρωτηθούμε αυτό τώρα με την αφορμή που έχουμε εδώ πέρα αυτές τις ε, γυναίκες που είναι πολεμιστές, είναι πολεμιστές για τον λαό τους, για το λαό όλου του Ιράκ και για όλες τις γυναίκες ε, που ήταν αυτόν τον αγώνα για όλη την ανθρωπότητα. Thank you. Last but not least, Εδώ είμαι. Ε, ευχαριστώ θερμά για το θάρρο σας. Απευθύνομαι στις δύο βραβευθύσες. Ε, σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για το θάρρο σας. θάρρος και προσωπικό θάρρος ε, ε, όλων των θυμάτων. Είναι πολύ σημαντικό να αναδείξει το βραβείο Ζαχάροφ τον αγώνα σας, ε, τα όσα υποφέρατε και να δείξουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. θα πρέπει να πιέσουμε ούτως ώστε κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη να προσφέρουν υποστήριξη και είμαι ευγνώμων στην κυρία Λόχ Μπίλερ να ε, καλέσουμε και την ε, τουρκική κυβέρνηση να βοηθήσει. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσουμε μάχη. Πολλά αφρικανικά ε, κράτη ε, έχουν ε, απογοητευτεί στον αγώνα τους. Ε, όμως η βράβευσή σας πιστεύω ότι θα δώσει ένα νέο έναυσμα ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία απέναντι σε όλες τις γυναίκες που βιάστηκαν και υποδουλώθηκαν. Νομίζω ότι ε, είστε ένα σύμβολο με το θάρρος σας απέναντι στη μάχη που οφείλουμε όλοι να δώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να βοηθήσουμε να και εμείς για να παραμείνετε δυνατές να σας στηρίξουμε. Είμαστε στο πλευρό σας και αν, έχ, δεν ξέρω, ε, αν έχετε κάτι να ζητήσετε ε, θα πρέπει να το κάνετε. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις η Νάντια ή η Λάμια. ممنون مش هر یکی شوی پیفتی و هر یکی که I would like to thank θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσοι μίλησαν και έδωσαν την άποψή τους. Whatever you all said, Πραγματικά, όπως είπατε όλοι σας, θα πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. E e e But these need to happen soon. Θα πρέπει όμως ε, αυτές οι προσπάθειες να γίνουν ε, γρήγορα, σύντομα, γιατί έχουμε κούρσα με το χρόνο και όσο περισσότερο χρόνο τριβούμε, τόσο θα αυξάνεται η αδικία εις βάρος του λαού μας. كهون مرة بسكنن كقواتا وقواتي بدمج أم كاربن جارك دي سلنجيت خب سكنو وبيض المصر عالم همو خطر يا داعش وفكرة داعش وإرهاب الوك داعش uh, It is very difficult for us. It's... Είναι πολύ δύσκολο για μας. Γι' αυτό και η υποστήριξή σας και η συμπεράστασή σας μας βοηθά να σταθούμε στα πόδια μας και να καταπολεμήσουμε τις θηριωδίες και τις βαναυσότητες που διαπράττονται εις βάρος μας. Ε,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 Ουδέποτε τα θύματα δεν θα φαντάζονταν ότι θα ερχόμασταν εδώ και θα μιλούσαμε μπροστά σε οποιαδήποτε βουλή ότι θα ακουγόταν η φωνή μας μετά τις μαζικές ε, θηριωδίες που υποστήκαμε. Πράγματα που μας ξεπερνούσαν, προβλήματα που μας ξεπερνούσαν. Ήρθαμε παρόλα αυτά γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Γι' αυτό ε, ζητούμε τη δική σας βοήθεια. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους θερμά που μιλήσατε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Και οι προτάσεις σας θα πρέπει να εφαρμοστούν τώρα, γιατί ο λαός μας ε, περιμένει εδώ και δύο χρόνια και δεν βαστάει άλλο πια. Και δεν είναι εύκολο να αντέξει ο κόσμο σε τέτοια κατάσταση και μάλιστα το έχει υποστεί δυόμιση χρόνια. We will not give up and we will continue. Δεν θα παραιτηθούμε πάντως, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και την εκστρατεία μας. Ε, ε, Um, και ελπίζω ότι και εσείς θα επιταχύνετε τις προσπάθειές σας για να δημιουργηθεί αυτή η ασφαλή ζώνη, γιατί ήδη είναι αργά. Αυτό που ήθελε το Ισλαμικό κράτος είναι να μας εξοντώσει, να μας εξολοθρεύσει να μας βύσει από το πρόσωπο της γης. Αλλά σας υπόσχομαι ότι δεν θα εγκαταλείψουμε, δεν θα παραιτηθούμε, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ευχαριστώ. Uh, Η κυρία Βαλενσιάνο, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε αυτό το τμήμα και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Τζαμίλεφ. Νομίζω ότι όλα τα είπαν και όλοι οι συναδελφοί εξέφρασαν την υποστήριξή τους που είναι και υποστήριξη τόσων Ευρωπαίων για την υπόθεση αυτή. Όλοι που βρισκόμαστε εδώ είμαστε εκπρόσωποι αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων Ευρωπαίων που βρίσκονται στο πλευρό σας. Οπότε είστε σίγουροι για κάτι τέτοιο και ελπίζω ότι αυτές τις μέρες θα το αισθανθείτε. Εμείς θα σας το δείξουμε όσο μπορούμε και θα συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή ούτως ώστε να απελευθερώσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά ζήτη. Um, Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια αυτά της υποστήριξης. Το βραβείο ε, απενεμήθη στις κυρίες. Η επιλογή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολο να διαλέξει κανείς ε, μεταξύ των υποψηφίων ο κύριος Τζαμίλεφ έδωσε μεγάλη μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το λαό του, για τη δικαιοσύνη. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και μπορείτε να μας απευθύνετε το λόγο. Ε, έχετε το λόγο αμέσως. Δραγέ Ναδία Μουράτ, Αγαπητή μου Νάντια Μουράντα, αγαπητή μου Λαμία Χατζή Μπασάρ, μέλη του Κοινοβουλίου. Όπως ε, είπατε, ήμουν μεταξύ των τελικών υποψηφίων για το βραβείο Ζαχάροφ, αλλά δυστυχώς στον κόσμο υπάρχει τόση ανομία, τόση αδικία ε, ακόμα και το γεγονός ότι ήμουν υποψήφιος και έφτασα μεταξύ των τριών, αυτό ήταν τεράστια ψυχολογική βοήθεια ε, για μένα και για τους Τατάρους της Κρυμαίας που χωρίς βία μέσα προσπαθούν να αντισταθούν στην ε, κατοχή της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Όταν είδα τον κατάλογο των υποψηφίων για το βραβείο θεώρησα ότι θα ήταν δίκαιο και θα ήταν μεγάλη ηθική υποστήριξη να ε, απονομηθεί στον Ελχάμο Τόρτε το βραβείο που καταδικάστηκε σε θάνατο από το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γιατί και εκείνος έδινε μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού του. Αλλά οι γενναίες αυτές οι γυναίκες, η Νάντια Μουράτ και η Λαμία Χατζή Μπασάρ, που αντιστάθηκαν στους εγκληματίες, στους ληστές αυτούς που ε, παριστάνουν τους ε, μουσουλμάνους και ε, κάνουν ζημιά στο Ισλάμ και τους μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο. Είμαι περήφανος για το βραβείο αυτό που πήρε το όνομά του από έναν ε, υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναν ε, ε, άνθρωπο που θεωρώ φίλο γιατί πολέμησε το σοβιετικό καθεστώς και υποστήριξε το λαό μου που μπόρεσε να επιστρέψει στην Κρυμαία και έσωσε και τη ζωή μου γιατί κατάφερε να με ελευθερώσει από τη φυλακή. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Ανδρέης Ζαχάροφ και είμαι πραγματικά ευτυχής που απενεμήθη στις ε, τόσο ε, θαραλές αυτές γυναίκες στο βραβείο. Νάντια Μουράντε, Λαμία Χατζή Μπασάρ, ε, σας παρακαλώ να θυμάστε πάντα ότι οι τρομοκράτες που διαπράττουν τα εγκλήματα αυτά δεν είναι μουσουλμάνοι. Ε, διαπράττουν εγκλήματα ενάντια και στους ίδιους τους μουσουλμάνους. Ευχαριστώ που είστε τόσο γενναίες, που είστε εν ζωή και που είστε εδώ μαζί μας. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Τζαμίλεφ που ήρθατε και που μας υπενθυμίσατε πως στο σημερινό μας κόσμο θα πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς τη δίνετε εδώ και χρόνια πολλά, γιατί έχουμε και παλινδρομήσεις δυστυχώς σε αυτόν τον αγώνα. Δεν έχει μείνει πολλή ώρα. Όποιο θέλει το λόγο, έχουν μείνει λίγα λεπτά. Αν κανείς έχει κάποιο σχόλιο να κάνει. Η, αντιπρο... η μας, η κυρία Σουίτσα. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Η Επιτροπή ε, για τη Συνεργασία με τη Ρωσία θα συνεδριάσει Τετάρτη, 2.30 με 4 παρατέταρτο. Και την Τρίτη θα συναντήσουμε ε, την αντιπροσωπεία της ε, κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας με την Τουρκία. 3.30 με 4.30 και θα συναντηθούμε με την αντιπροσωπεία του Ιράκ. Η συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη, 4 με 5,5. Και στη συνεδρίαση αυτή ε, για το Ιράκ ε, θα είναι παρούσες και και την ε, Τρίτη και Τετάρτη στι συναντήσει για τη Ρωσία και την Τουρκία θα έχουμε χρόνο και για ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ντουντάρ, Τζαν Ντουντάρ και με τον κύριο Τζαμίλεφ. Οπότε όσοι δεν είχατε την ευκαιρία σήμερα ή το χρόνο να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας θα έχετε ε, στη συνεδριάση των δύο αντιπροσωπείων για τη σχέση με την Τουρκία και τη Ρωσία την ευκαιρία να το κάνετε. Ωραία. Ε, έχει προχωρήσει η ώρα και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν και στις συνεδριάσεις ε, της Επιτροπής ΑΦΕΤ και των ε, σχετικών αντιπροσωπιών ε, και της αντιπροσωπίας με το Ιράκ να συναντηθείτε με τους φιναλίστ και τις βραβευθύσεις. Είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Για... Μιλήσετε για ανθρωπιστική υποστήριξη που χρειάζεται και συνδρομή για την κοινότητά σας. Εμείς είμαστε αρμόδιοι στη δική μου επιτροπή για το θέμα αυτό, οπότε θα πρέπει με τα άλλα μέλη της Επιτροπή ανάπτυξη να προωθήσουμε αυτό το θέμα τη ανθρωπιστική συνδρομή προ την κοινότητα για ζητή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συνθήκε διαβίωση των προσφύγων στην Ελλάδα, εγώ και ο κύριος Γκερέρο, που είναι ο μόνιμος ηγετής για την ανθρωπιστική βοήθεια, έχουμε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκε διαβίωση των προσφύγων ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Και αναφερθήκατε κι εσείς, ε, Λάμια, για την έλλειψη πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση και αυτό είναι προτεραιότητα της Επιτροπής μας και θα το φροντίσουμε, θα το εξετάσουμε τουλάχιστον. Οπότε θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συναντηθούμε με τις βραβευθύσεις. Αύριο θα γίνει η, απονομή, η πανηγυρική απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Θα είμαστε όλοι στην Ολομέλεια για την τελετή και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και τη συμπαράστασή μας προς τις βραβευθύσεις και προς το λαό ZD. Και φυσικά δεν σταματούμε εδώ, δεν σταματούμε με το βραβείο. Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους βραβευθέντες. Πέρσι είχαμε την ε, ε, την απονομή στον ε, ε, φυλακισμένο από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζουμε την επαφή με την οικογένειά του, με τους δικηγόρους του και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Αυτό θα ήθελα να πω από τον κύριο Τζεμίλεφ προς την Άντια και τη Λάμια, ότι είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε όχι μόνο με την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ, αλλά και τη μέρα μετά από αυτό και στη συνέχεια και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία και την εβδομάδα αυτή αλλά και στο μέλλον για να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη και για το λαό σας που τον αξίζει και για τον λαό των Τατάρων που επίσης το αξίζουν.